Now I give. Okay, we are going to start the vote. If you are so kind to take your seats. Προκειμένου να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες, παρακαλώ να καθίσετε. To present a point of order. Υπάρχει έτοιμα από την κυρία Ρέγνερ. Κυρία Ρέγνερ, έχετε το λόγο. Danke schön, Herr Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπάθησα στην προηγούμενη συζήτηση για την ανάπτυξη να σηκώσω μπλε κάρτα ε, απευθυνόμενη προς τον κύριο Ούμπεμαϊα αλλά ε, δεν μπόρεσα γιατί μόλις μίλησε εξαφανίστηκε μετά έφυγε μέσα από την αίθουσα γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να παρακαλέσω οι ευρωβουλευτές να παραμένουν με στην αίθουσα για λίγο έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να τους υψώσει μπλε κάρτα να έχει έστω αυτή την ευκαιρία